Ο πρόεδρος έλαβε ένα νέο διορισμό από πλευρά σοσιαλιστών που θα καταγραφεί στα πρακτικά. Μιλάμε ότι για την αντικατάσταση της κυρίας Στάινρουκ από τον κύριο Αρν Κον ε, σε σχέση, στην ε, αντιπροσωπεία σχέσεων